Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο πραγματικά είναι πολύ δραστήριο σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, σε ευχαριστώ. Θα κλείσω εδώ τη συζήτηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση των Ρωμά στα κράτη-μέλη. Θα συνεχίσουμε την ε, εργασία μας, με βάση, τις εργασίες μας με βάση την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εκείνους που θα κάνουν ε, παρεμβάσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Δεν θα υπάρξουν αυθόρμητες παρεμβάσεις για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καταρχάς, θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Βασιλείου, η οποία θα μας παρουσιάσει την δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή της Αντιπροέδρου και της ΥΠΑ της Εκπροσώπου της Ένωσης. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν τη δήλωση Άστον για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς. Εκ μέρους της είπα της εκπροσώπου Κάθη Άστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα των πυρομαχικών διασποράς μαζί σας σε μια τόσο επίκαιρη χρονική στιγμή όπου διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ για να απαγορεύσουμε αυτά τα τρομερά όπλα σε παγκόσμια κλίμακα επιτέλους. Τον Ιούλιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε την θέση σε ισχύ της σύμβασης για τα πυρομαχικά διαποράς ε, την 1η Αυγούστου του 2010. Εν συνεχεία, τον Νοέμβριο του 2010, η πρώτη συνάντηση των χωρών έλαβε χώρα στο Λάος και συγκεκριμένα ε, υιοθετήθηκε ένα σχέδιο δράσης στη Βιεντιάν. Αυτό ήταν ένα αξιέπαινο πρώτο βήμα για να υποστηρίξουμε την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς και στην συνάντηση της Βιεντιάν πέρυσι και στη δεύτερη συνάντηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2011 στη Βηρητό φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας ένθερμος υποστηρικτής των διεθνών προσπαθειών για να αντιμετωπίσουμε το φοβερό ανθρωπιστικό πρόβλημα και τις φοβερές ανησυχίες που θέτουν τα πυρομαχικά αυτά διασποράς. Σήμερα, 66 κράτη είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς. 108 κράτη έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος σε, ε, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα για να συμπεριλάβουμε τους μεγαλύτερους παρασκευαστέ τέτοιων πυρομαχικών στο, στη συνολική προσπάθεια που κάνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση ό,τι αφορά αυτά τα πυρομαχικά. Δυστυχώ, φέτο αποδείχτηκε ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι φανταζόμαστε. Η ύπατη εκπρόσωπος ανησυχεί τα μάλα για τη χρήση τέτοιων πυρομαχικών διασποράς εναντίον άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη και ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις του Μουαμάρ Κανταφή να μην χρησιμοποιήσουν τέτοια πυρομαχικά εναντίον αμάχων. Ούτε πυρομαχικά διασποράς βεβαίως, ούτε άλλα όπλα όλα τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε οι άμαχοι να προστατευθούν από τις επιπτώσεις τέτοιων πυρομαχικών. Και τα μη εκραγέντα ε, κομμάτια τέτοιων πυρομαχικών δια, ε, διασποράς. Αυτή τη βδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο ε, για τα πυρομαχικά αυτά στη Γενέβη στο πλαίσιο της ε, διάσκεψης για την μεταρρύθμιση της σύμβασης κάποιων ε, συμβατικών όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει στεναρά ότι οποιοδήποτε νέο μέσο πρέπει να σεβαστεί τους στόχους της ενίσχυσης της του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Η ύπατη εκπρόσωπος και εγώ σημειώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή στο ψήφισμα του 2008 και το 2010 και ξανά το 2011 κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς ε, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο και χωρίς να παρακάμψουν την σύμβαση υιοθετώντα εγκρίνοντας ή επικυρώνοντας το πρωτόκολλο 6 CCW για την χρήση των πυρομαχικών διασποράς που δεν θα είναι συμβατό με την απαγόρευση της χρήσης τέτοιων πυρομαχικών με βάση τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς. Πιστεύουμε στεναρά ότι σε ό,τι αφορά τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για ένα πρωτόκολλο CCW για τα πυρομαχικά διασποράς, τέτοιες διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν σε ουσιαστικές βελτιώσεις επιτόπου, λαμβάνοντας υπόψη και τα ανθρωπιστικά θέματα και τα στρατιωτικά θέματα, που πρέπει να είναι συμβατά και συμπληρωματικά με τα όσα προβλέπει η Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς. Πιστεύουμε ότι αυτό το εργαλείο θα έχει και διατάξεις για τη συνεργασία και τη βοήθεια και ότι θα αποτελέσει σημαντική ανθρωπιστική συμβολή προβλέποντας άμεση απαγόρευση για τη χρήση, την παραγωγή, τη μεταφορά των πυρομαχικών διασποράς. Αυτό θα επιτρέψει την διεθνή κοινότητα να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς σωστή κατεύθυνση και να πλησιάσει στο σκοπό που είναι ανθρωπιστικός. Σε ό,τι αφορά αυτό τον ε, τελικό μας σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει και αυτή και να συνεισφέρει στο βαθμό που μπορεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ε, σε αυτό το σημαντικό έργο, ούτω ώστε να ενισχύσει τη σημασία της CCW, τη σύμβαση δηλαδή για τα συμβατικά όπλα, και να ενισχύσει το κανόνα ότι τα δεν μπορούν τα, μέλη να επιλέγουν ε, τα όπλα τους ε, με όποιον τρόπο θέλουν, χωρίς κανένα φραγμό. Τα πυρομαχικά διασπορά είναι αντίον ε, διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις τους ε, στον άμαχο πληθυσμό με όλα τα απαραίτητα μέσα. Παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο για να υλοποιηθούν οι ανθρωπιστικοί στόχοι της Σύμβασης των πυρομαχικών διασποράς μέσω αποτελεσματικής παροχής βοήθειας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιτόπου, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, των τη βοήθεια των θυμάτων ε, ναρκών ή πυρομαχικών διασποράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει καμία διάκριση. Πρέπει να σεβαστούμε πλήρως τις υποχρεώσεις της Σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς και αυτό θα είναι βαθύτατη πρόκληση για πολλά συμβαλόμενα κράτη ανά τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει το περίπλοκο του θέματος και είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια σε κράτη στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τα εθνικά τους προγράμματα με αποτελεσματικό τρόπο, να σεβαστούν τη σύμβαση και να εξασφαλίσουν συνέργειες με άλλα εξίσου σημαντικά διεθνή εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά δεσμευμένη στην προσπάθεια σεβασμού των νομικών υποχρεώσεων της ε, Σύμβασης και της μετατροπής αυτών των νομικών υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά τη συζήτηση τώρα, θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και καταρχήν θα δώσω το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ στον κύριο Γκάλερ για δύο λεπτά, για μισή λεπτά. Παρακαλώ. Είναι καλό που το κοινοβούλιο μας στο πλαίσιο αυτού του ψηφίσματος ε, όσον αφορά την αναθεώρηση της σύμβασης τη Σύμβαση για τα ορισμένα συμβατικά όπλα ασχολείται με το ζήτημα των πυρομαχικών διασποράς. Το κείμενο θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια περαιτέρω συμβολή του Κοινοβουλίου για την εξέλιξη των ανθρωπιστικών μας προσπαθειών όσον αφορά τον έλεγχο των πυρομαχικών αυτών. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο βασικά αιτήματα. Ε, πρώτον, ε, να τηρηθεί η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς. Ε, θα ήθελα καταρχήν να αναπτύξω το στατιωτικό επιχείρημα έναντι του πολιτικού ανθρωπιστικού επιχειρήματος. Όσον αφορά την ε, αποστατική άποψη, τα πυρομαχικά διασποράς είναι από τα πιο ε, αποτελεσματικά συμβατικά όπλα. Ε, γίνεται σε δρόμους ή σε σημαντικές υποδομές εν γέννη. Αυτή είναι η καθαρά στρατιωτική πτυχή η οποία διαφοροποιείται από την ανθρωπιστική ε, πτυχή. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς. Το ολέθριο εδώ είναι ότι η χρήση πολύ συχνά ε, γίνεται με, με έναν τρόπο που είναι εξαιρετικά βλαβερός για την ανθρώπινη ζωή. Ε, είναι πολύ ψηλά αυτά τα ποσοστά ανθρώπινων θυμάτων τυφλών θυμάτων ε, και αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Λιβύη γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα από τον Καντάφη και είναι μια ξεκάθαρη απειλή του πληθυσμού σε καταστάσεις ένοπλης σύραξης. Η ανθρωπιστική απειλή ε, μπορεί να αποτελέσει μία υποθήκη ε, έναντι μιας, σε σχέση με μία δυνατότητα ανοικοδόμησης της χώρας. Γι' αυτό θα πρέπει να απαγορευτούν αυτά τα πυρομαχικά διασποράς και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σχετικές προσπάθειες. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει κάνει ενισχυμένες ε, προσπάθειες να υποστηρίξει τις τρίτες ε, χώρες για να καταστρέψουν τα αποθέματα των πυρομαχικών διασποράς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλερ και τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Κουαλτιέρη. Πρόεδρε, όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, αυτά τα πυρομαχικά διασποράς είναι ένα εργαλείο θανάτου για τον άμαχο πληθυσμό και επομένως πρέπει να τα απαγορεύσουμε για λόγου πολιτισμού. Ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση εδώ και καιρό. Η θέση σε ισχύ της σύμβαση του Όσλο ήταν μια σημαντική επιτυχία. Αλλά σήμερα λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, από τη θέση, ε, ένα ισχύ ε, βλέπουμε ότι γίνεται μια σημαντική και περίπλοκη απόπειρα να την αποδυναμώσουμε με, αυτό το, με το πρόσθετο πρωτόκολλο ε, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Γενέβη, το οποίο θα νομοποιούν νομιμοποιούσε την χρήση αυτών των βομβών ε, διασποράς. Αυτό το πρωτόκολλο δεν πρέπει να υπογραφεί από αυτούς που είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης του Όσλο. Γιατί όπως υπόθηκε και από την ίδια την Επίτροπο είναι σε άμεση αντίφαση με την ίδια τη Σύμβαση. Ε, και θα ξεκίναγε μία, ένας φαύλος κύκλος και για τις άλλες χώρες που θέλουν να συνεχίσουν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα όπλα. Και επίσης θα δημιουργούσε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο σε διεθνές επίπεδο. Το επιχείρημα ότι το πρωτόκολλο θα βελτίωνε την κατάσταση γιατί θα υπογραφόταν από χώρες που δεν πρόκειται να υπογράψουν τη σύμβαση του Όσλο μας φαίνεται απίστευτο και θα θέλαμε ε, να ακούσουμε την άποψη της είπα της εκπροσώπου Άστον. Θα θέλαμε να, να την ακούσουμε να εκφράζεται ε, με καθόλου αμφίσιμα λόγια, με σαφή λόγια. Γιατί νομίζω ότι θα δυναμίτιζε αυτό το πρωτόκολλο την ίδια την ε, σύμβαση ε, για τη χρήση των πυρομαχικών διασποράς που έχουν παραχθεί μετά το 1980 που είναι τα περισσότερα. Επιτρέπει μια τεράστια περίοδο μεταβατική και ούτω ή άλλω μην ξεχνάτε ότι αυτά τα πυρομαχικά είναι πολύ επικίνδυνα για του άμαχου και δεν ε, θέτει στόχου για την καταστροφή των αποθεμάτων των κρατών. Επομένω είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να μην υποστηρίσουν τη θέση σε ισχύ αυτού του πρωτοκόλου και είπα ότι εκπρόσωπο να δεσμευτεί ούτω ώστε όλε οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν μια σαφή στάση και ενιαία στάση υπέρ της ε, οριστικής απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς. Ε, το κοινό ψήφισμα, επομένως, που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα και πιστεύουμε ότι θα ε, εγκριθεί από μια ευρεία πλειοψηφία εν το συνόλο του. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάκε για δύο λεπτά εκ μέρους των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων. Ε... Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με τους προηγούμενους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα για αυτό το κοινό ψήφισμα. Η Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς τέθηκε σε σχέση το 2010 και συμπερέλαβε τις περισσότερες χώρες μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να παραγωγηθούν τα πυρομαχικά διασποράς γιατί δημιουργεί ολέθριες βλάβες στον άμαχο πληθυσμό. Από μια ανθρωπιστική πλευρά πρόκειται για πραγματική καταστροφή. Αλλά ορισμένες χώρες μέλη δυστυχώς πιστεύουν ότι τα πυρομαχικά διασποράς είναι σημαντικά για την ασφάλεια και την οικονομία τους. Τώρα, δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω τη σημασία της ασφάλειας, αλλά υπάρχουν πιο εκλεπτευσμένοι και λιγότερο επιζήμιοι τρόποι για να την εξασφαλίσει κανεί. Πέρα από τη χρήση υπάρχει βεβαίω και το εμπόριο. Πρόσφατα ακούσαμε εκθέσεις για τη χρήση προμαχικών διασπορά στη Λιβύη και προφανώ ορισμένε χώρε μέλη συμμετείχαν στην ε, πώληση αυτών των όπλων. Ε, θα υπάρξει μια συζήτηση για το πρωτόκολλο 6 για μια, ε, κατά τη διάρκεια μια σύμβαση αναθεώρηση ε, τη σύμβαση για τα συμβατικά όπλα και δεν είναι συμβατή με τι δεσμεύσει που έκαναν οι χώρε μέλη. Αντιθέτω, αντί να υπονομεύσουμε ε, τη σύμβαση για τα πυρομαχικά διασπορά θέλουμε περισσότερα μέλη να την προσυπογράψουν. Θα προσχωρήσουν χώρες που δεν θέλουν να παράγουν ή να αποθηκεύουν όλα τα πυρομαχικά διασπορά ή θα δεσμευτούν ε, ε, στην απαγόρευση τέτοιου είδου δραστηριοτήτων. η να αποθηκευουν ολα τα πυρομαχικα διασπορα η θα δεσμευτουν στην απαγορευση τετοιου ειδου δραστηριοτητων Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε μια συνολική απαγόρευση των πυρομαχικών διασπορά. Και αν θέλουμε να διανοηθήσουμε εδώ έναν ενεργό ρόλο, θα πρέπει να δώσουμε το σωστό παράδειγμα, συμπεριλαμβάνοντα όλε τι χώρε μέλη ανεξαιρέτω. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ πολύ με τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο προηγούμενα. Τα πυρομαχικά διασποράς είναι πάρα πολύ σκληρά, επικίνδυνα ε, πυρομαχικά. Φανταστείτε ένα παιδί να πάει να πιάσει ένα τέτοιο αντικείμενο και που εκρήγνεται και το παιδί αυτό ε, διαμελίζεται. Ένα τρίτο των θυμάτων είναι παιδιά Πάρα πολλοί τραυματίζονται όταν ακολουθούν κανονικέ δραστηριότητε τη καθημερινή ζωή, όπω συμβαίνει στη Λιβύα. Πολλοί από εμά, ε, ευρωβουλευτέ, ε, η κοινωνία των πολιτών, όλοι προσπαθήσαμε να υπογραφεί η σύμβαση του Όσλο του 2008 κατά των πυρομαχικών διασπορά. Αυτή η απαγόρευση διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώ σήμερα στη Γενέβη, στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών ε, για αυτό το θέμα, Κάποιοι θέλουν να καταψηφίσουν τη σύμβαση σε σχέση με το πρωτόκολλο 6 και θέλουν να καταψηφίσουν ανθρωπιστική νομοθεσία διεθνούς χαρακτήρα. Δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και την ύπατη εκπρόσωπο για τον σαφή τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν σήμερα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συμφώνησαν σε ένα πολύ καλό ψήφισμα και σε στενή συνεργασία που είχαμε όλοι μεταξύ μας των λεχθέντων είμαι πεισμένη ότι με ενωμένη φωνή οι Ευρωβουλευτέ, το Ευρωκοινοβούλιο, αποκοινούμε την εκπρόσωπό μα για τα εξωτερικά, κάθε άστον, θα εισακουστούμε στη Γενέβη από αυτού που έχουν υπογράψει και από αυτού που ε, θα επικυρώσουν και εκείνου που δεν έχουν υπογράψει κατά αυτών των πυρομαχικών διασπορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στη συνέχεια εξ ονόματος ε, της ομάδας Ενωτικής Αριστεράς. Η κυρία Λόσενγκ θα λάβει τον λόγο 1,5 λεπτό. Χαιρετίζω εξ ονόματος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ενωτικής Αριστεράς ε, την πολύ καλή διακομματική συνεργασία που είχαμε και την πλειοψηφική υποστήριξη του κοινού ψηφίσματος κατά της χρήσης βομβών διασποράς και πυρομαχικών διασποράς. Είναι σημαντικό αυτό το ψήφισμα και σημαντικό μήνυμα στον αγώνα κατά αυτών των δολοφονικών όπλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πυρομαχικά διασποράς και οι βόμβες στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν παντού εκεί χρησιμοποιήθηκαν και μάλιστα υπενθυμίζω στο Ευρωκοινοβούλιο και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα, να αποθηκεύονται, να διατηρούνται ή να παράγονται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε για την άμυνα ούτε για την διασφάλιση συνόρων απευθύνω κατεπηγόντως έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη το προτινόμενο κείμενο του έκτου πρωτοκόλου για τα πυρομαχικά διασποράσα και για την απαγόρευση αυτών των όπλων να μην υποστηρίξουν το κείμενο αυτό. Το κείμενο αυτό απαγορεύει και δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό τις βόμβες που είχαν χρησιμοποιηθεί, είχαν παραχθεί πριν από, ε, στο παρελθόν ήδη. Αυτό σημαίνει ότι οι, ε, μέχρι σήμερα παραγόμενε βόμβε επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται περαιτέρω. Δεν μπορούμε όμω να δεχθούμε κάτι τέτοιο με κανένα τρόπο. Η Σύμβαση για την Απαγόρευση των Πυρομαχικών Διασπορά, που τον Αύγουστο 2010 άρχισε να ισχύει απαγορεύει όλων των ειδών ε, πυρομαχικά διασπορά και βόμβε. και αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονα με τον οποίο θα μετρήσουμε Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος τώρα, κυρίες και κύριοι, των παρεμβάσεων των Ευρωβουλευτών και πάλι θα λάβει τον λόγο λοιπόν στη συνέχεια η κυρία Επίτροπος, η κυρία Βασιλείου παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωβουλευτές για τη συνεισφορά τους και για το ότι μας δίνουν την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το κρίσιμο θέμα για να αντιμετωπίσουμε το καυτό ανθρωπιστικό πρόβλημα που θέτουν τα πυρομαχικά διασποράς. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τη δέσμευσή της για να επιτευχθεί μια παγόρευση σε αυτά τα πυρομαχικά μέσω ενεργούς πολιτικής δράσης ε, και σε επίπεδο σύμβασης και σε ε, σε επίπεδο συμβάσεων, ε, τη σύμβασης μάλλον για τα συμβατικά όπλα. Θέλω να εκφράσω τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αυξήσουμε τον αριθμό των υπογραφών και επικυρώσεων και οι φιλοδοξίες μας να γίνουν πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να δίνει διεθνή βοήθεια και συνεργασία απλουστεύοντας τις δραστηριότητες εναντίον των πυρομαχικών διαφοράς, διασποράς στις πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει τι περίπλοκο είναι το ζήτημα αυτό ε, και η εφαρμογή της ε, σύμβασης για τα συμβατικά όπλα και το σχέδιο δράσης της Βιεντιάν ε, απαιτούν και οικονομικούς πόρους αλλά και πολιτική δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει τα κράτη προς αυτή την προσπάθεια. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημείου στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε έξι ψηφίσματα.